Έρχεται η συνεδρίαση. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση της κυρίας Ζολή. Δεύτερη αναθεώρηση Συμφωνίας Εταιρικής σχέση και Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Συμφωνία Κοτονού. Ο πρώτος ομιλητής, η πρώτη ομιλήτρια μάλλον, διορθώνει ο πρόεδρος, εάν είναι παρούσα, είναι η κυρία Εύα Ζολή. Jolly, are you ready? Είστε έτοιμοι κυρία Ζολή. Έχετε το λόγο. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire et chers collègues. Κύριε Πρόεδρε, η Επίτροπη, αγαπητοί συνάδελφοι, η αναθόρεση της Συμφωνίας Κοτονού μας ε, βοηθάει να μάθουμε κάτι από τις κρίσεις, την οικονομική, την χρηματοοικονομική, την κοινωνική, την επιτιστική, την αλλαγή του κλίματος, τις προκλήσεις ε, στον τομέα της ενέργειας, η επιμονή της φτώχειας, μοντέλα τα οποία έδειξαν ότι η σημερινή μας αντιμετώπιση έχει τα όρια της και ότι η κρίση είναι πολυδιάστατη. Η έκθεση την οποία σας υποβάλλουμε σήμερα υιοθετήθηκε ομόφωνα από την Επιτροπή Ανάπτυξης και είναι κατά κάποιο τρόπο ένα πρώτο βήμα σε αυτή την απαραίτητη αναθεώρηση. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συνεκτικοί στην απάντησή μας. Η εμπορική πολιτική, η αλία και η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να έχουν συνοχή έτσι ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη, καταπολέμηση της φτώχειας και καλύτερα εισοδήματα για όλους. Δυστυχώς αυτό σήμερα δεν συμβαίνει και λυπούμε πολύ γι' αυτό. Το εμπόριο είναι αυτό σκοπό σήμερα και όχι μέσο για την αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτόν τον τρόπο θυσιάζουμε τους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών προς όφελος των πολυεθνικών. Οι εταιρικέ σχέσεις και οι συμφωνίες σήμερα λοιπόν αφισβητούνται από τις χώρες ΑΚΕ και τις κυβερνήσεις τους και την ίδια ώρα υπάρχει η αντιμετώπιση τους ως απειλή για τις οικονομίες τους. Σήμερα το θέμα της γεωργίας είναι το πιο προβληματικό και είναι εγκαταλελειμμένο θέμα ως προς τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χώρες ΑΚΕ. Πάνω από το 60% του πληθυσμού των χωρών αυτών ζουν από τη γεωργία και στην Ήπεθρο. Την ίδια ώρα βλέπουμε ότι τα εισοδήματα από αυτόν τον τομέα είναι ελάχιστα και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την φτώχεια χωρίς να υπάρξει επισητιστική επάρκεια και αυτάρκεια. Και θα πρέπει λοιπόν η ανάπτυξη να μπει στην καρδιά της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εταιρική σχέση με τους αγρότες, με τους γεωργούς αυτών των χωρών να διασφαλίσουμε την επιστημιστική τους ε, ασφάλεια. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα νέο φαινόμενο που απειλεί τις χώρες αυτές. Είναι η κατάχρηση των ε, καλλιεργήσιμων περιοχών από εξωτερικούς φορείς. Η Κίνα, το Κατάρι, η Σαουδική Αραβία κατέχουν σήμερα χιλιάδες ε, στρέμματα στις χώρες αυτές. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθεί με το θέμα αυτό έτσι ώστε να αποφευχθούν εξεγέρσεις και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αγαθά όπως τη γη και το νερό σαν αναφέρετα δικαιώματα αυτών των πληθυσμών. Και ένα άλλο θέμα που μου φαίνεται πολύ σημαντικό είναι η φορολογική παράδειση. Καθότι οι συνέπειες της ύπαρξης αυτών των φορολογικών παραδείσων είναι πλήγματα για τις χώρες αυτές και τις οικονομίες τους. Σήμερα παράνομες χρηματοοικονομικές ροές ξεπερνούν το δεκαπλάσιο της επιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι θέμα αξιοπιστίας και ένα πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η συμφωνία, η υπογραφή μιας δεσμευτικής συμφωνίας για τις πολυεθνικές, έτσι ώστε να αναγκάζονται να δηλώνουν τα κέρδη τους και τον κύκλο εργασιών τους σε όλες τις χώρες τις οποίες είναι παρούσες, έτσι ώστε να αποφευθούν αυτές οι καταχρήσεις για την οικονομία των αναπτυσσόμενων χωρών. Επίσης το δημοκρατικό έλλειμμα, κάτι το οποίο δεν απασχόλησε μέχρι τώρα τα κοινοβουλιά μας. Η κοινοβουλευτική συνέλευση ίσης εκπροσώπησης θα πρέπει να ενισχυθεί για αυτό το σκοπό κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ελπίζω αυτοί οι οποίοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις να αναλάβουν με σθένος την αναθεώρηση αυτής της συμφωνίας έτσι ώστε να υπογραφεί μια αναθεώρηση προς όφερος των χωρών ΑΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, Ευρωβουλευτές, η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, της οποία είμαι πρόεδρος, αποφάσισε να λάβει θέση σχετικά με την αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού που έχει ήδη ξεκινήσει για δύο λόγους. Πρώτον, διότι οι εμπορικές συναλλαγές αποτελούν ουσιαστικό μέρος των σχέσεων μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και κατά δεύτερο λόγο, επειδή αυτή η Συμφωνία του Κοτονού καθιέρωσε σχέσεις, εταιρικές σχέσεις οικονομικές βάσει συμφωνιών που είναι καθαρά ουσιαστικά εμπορικές. Γι' αυτό αποφασίσαμε να παρέμβουμε υποβάλλοντας μία έκθεση για την οποία είμαι εγώ υπεύθυνο. Στην έκθεση αυτή εκφράζουμε δύο ανησυχίε. Πρώτον, την ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι ιδιαιτερότητες των συμφωνιών αυτών και κατόπιν πρέπει να τηρούνται ήδη υπάρχουν συμφωνίες και να διαπιστωθούν οι συνέργειες που θα <clears throat> που υπάρχουν, που έχουν ήδη διαμορφωθεί και να προστατευθούν. Οι χώρες και πρέπει λοιπόν όλοι οι ενδιαφερόμενοι να προασπίσουν αυτές τις ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Ο κύριος Δεγκούχτ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτιμώ ιδιαίτερο το ενδιαφέρον που δείχνεται για τη δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού και μάλιστα με μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης που ε, μας δίνει και μεγάλη ανάλυση επί του θέματος. Σε όλη τη διαδικασία προτεραιότητά μας είναι να ενημερώνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπως κάναμε και τους προηγούμενους μήνες. Οι διαπραγματεύσεις ε, έχουν ε, ε, βρει την κατάλληλη ορμή και έχουν πλέον ενταχθεί στην τελική φάση. Η τελευταία κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση θα δείξει ακριβώς ότι έχουμε φτάσει προς το τέλος. Προβλέπεται και το Μάρτιο μια κοινή υπουργική διάσκεψη βάσει και τη Συμφωνία Κοτονού. Θα ήθελα τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις επί της εκθέσεως ε, η έκθεση είναι ιδιαίτερο χρήσιμη διότι μπορούμε να λάβουμε υπόψη κάποιες θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να σας πω αναφορικά την ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ των ε, Κοινοβουλίων Χωρών ΑΚΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό επιβεβαιώνει τη θέση μας, όπως επίσης και τη σημασία που έχετε προσδώσει στην αλλαγή του κλέματος, κάτι το οποίο συμμεριζόμαστε και εμείς και αυτό θα προκύψει και στο τελικό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να εστιάσω σε τέσσερα θέματα, τα οποία βασίζονται στη σημασία της κοινοβουλευτικής διάστασης ε, στην κοινή ε, κοινοβουλευτική συνέλευση. Η έκθεση προσδίδει ιδιαίτερα σημασία σε αυτό. Θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση στη Συμφωνία Κοτονού από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένω, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να αποδυναμώσουμε την κοινοβουλευτική συνέλευση. Ε, ίσα ίσα θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία βάσει των υφιστάμενων και των μελλοντικών ε, συμφωνιών οικονομική και εταιρική σχέση και ε, κοινών συμφωνιών. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τους θεσμούς και με τους κοινοβουλευτικούς φορείς των χωρών ΑΚΕ. Σε αυτό λοιπόν το αναδεόμενο ε, περιβάλλον η μείωση των ε, ολομελιών ναι μεν είναι λογική αλλά αυτό θα πρέπει να συμφωνηθεί και με όσους ενδιαφέρονται περισσότερο επί του θέματος και είναι διατεθειμένη να επανεξετάσει τη θέση της. Θα θέλαμε να μάθουμε και κάποια περισσότερα πράγματα από το Κοινοβούλιο. Πώς βλέπετε ε, το θέμα αυτό της πολιτικής και θεσμικής ανταλλαγής απόψεων. Επίσης, δεν υπάρχει μόνο ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ε, συνέργεια μεταξύ ημών και των θεσμικών οργάνων της Συμφωνίας Κοτονού, αλλά και ε, να δούμε κατά πόσον γίνονται σεβαστές οι διατάξεις της Συμφωνίας Κοτονού, διότι το καθεστώς εμπορίου είναι πλέον παροχημένο. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις περιφερειακό, στις ε, περιφερειακές συμφωνίες εταιρικής σχέσης, και εδώ η Επιτροπή Ανάπτυξης λέει ότι δεν είναι πολιτικά επιθυμητό ούτε δυνατό να υπάρχουν μονομερεί ε, καθεστώτα εμπορίου όπως το ESP και το ESP sin στη Συμφωνία Σκοτονού διότι αυτό εξαρτάται από αυτόνομα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιθέτως, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε θέματα εμπορίου και ανάπτυξης εν γέννη και να βοηθήσουν τα θέματα εμπορίου. Στη νέα συμφωνία εκφράζεται την ανησυχία ότι θα αυξηθεί η περιφερειακή διάσταση, κάτι το οποίο μπορεί να αποδυναμώσει τη συνοχή της ομάδας ε, ΑΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η περιφερειακή διαφοροποίηση είναι ευκαιρία και όχι απειλή. Η περιφερειακή ε, ολοκλήρωση είναι θεμελιώδης σημασία για τις χώρες ΑΚΕ και αυτή η πραγματικότητα θα πρέπει να ενσωματωθεί στη Συμφωνία Κοτονού για να μπορέσουν να υλοποιήσουν και τους στόχους που έχουν αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα διαταραχθεί η ομάδα των χωρών ΑΚΕ και ε, θεωρούμε ότι είναι η σωστή προσέγγιση. Να αναφερθώ τώρα σε κάποια σημεία τα οποία επισημαίνεται στην έκθεσή σας. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η αλλαγή του κλίματος ε, ε, και οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια που αναφέρονται και στην παρούσα διαδικασία. Επίση, μα ενδιαφέρει το θέμα τη επιστημιστική ασφάλεια ε, στην περιφερειακή διάσταση και μα ενδιαφέρει και η καλή, η χρηστή διακυβέρνηση. Η χρηστή διακυβέρνηση είναι θεμελιώδη αρχή τη Συμφωνία Κοτονού και ξεκινάει από το άρθρο 9 της συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει του άρθρου 9 ετοιμάζει μια νέα πρόταση ε, για την ε, αναπτυξιακή συνεργασία και θέλει να προωθήσει περαιτέρω αυτές τις πτυχές ε, στη νέα διαδικασία αναθεώρησης. Θεωρώ λοιπόν ότι συμμεριζόμαστε τον ίδιο στόχο, θέλουμε να έχουμε θεμετό ε, αποτελεσματικά φορολογικά συστήματα και αποτελεσματικές φορολογικές διοικήσεις, καθώς επίσης και την ενίσχυση της ε, συμμετοχής των αναπτυσσόμενων χωρών στη φορολογική διαδικασία. Επίσης, ε, λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαβουλεύθηκε με μια μεγάλη σειρά φορέων πριν ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης, παράγραφος 2, σημείο 8. Συμφωνώ απολύτω ότι για το μέλλον των σχέσεων χωρών και Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020 χρειάζεται μια κοινή διαδικασία διαβούλευση, ίσω υπό τη μορφή πράσινη βίβλου. Θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα τη παρούσα διαδικασία αναθεώρηση και θα αυτά θα αποτελέσουν τη βάση ε, των όσων θα μάθουμε για το μέλλον. Ο κύριος Πρέντα για δύο λεπτά. Πρώτα θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ζολή, κύριε Πρόεδρε, για την έκθεση αυτή. Τα θέματα τα οποία περιέχει είναι ιδιαίτερα σημαντικά προκειμένου να εξασφαλίσουν να αποτελέσει η Συμφωνία του Κοτονού τη βάση των σχέσεων με τις χώρες ΕΚΕ αξιόπιστο μέσο στα πλαίσια της διαμόρφωσης ε, των νέων συνθήκων. Οι διαπραγματεύσεις ε, γίνονται σε μια δύσκολη στιγμή. Οι χώρε εκεί έχουν επηρεαστεί έντονα από την οικονομική κρίση και την επισητιστική ανασφάλεια και την κλιματική αλλαγή. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η θεσμική πρόκληση για όλε τι φάσει των διαπραγματεύσεων. Σκοπό είναι να εκφράζονται σαφώ η τάση της περιφερειοποίηση των σχέσεων μεταξύ των χωρών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το αναθεωρημένο κείμενο πρέπει να περιέχει όλα τα περτούμενα συστατικά, πρέπει να το φροντίσουμε αυτό για αποτελεσματική συνεργασία που θα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι εξ ονόματος του ΕΛΚ έχω καταθέσει πέντε τροπολογίες οι οποίες κατά την άποψή μου επιτρέπουν να, καλύτερη ανάγνωση των διαφόρων σημείων. Σχετικά με το σημείο 29 πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα της κυριότητας της κατοχής αρωτρέων εκτάσεων. Και οι πολυεθνικές εταιρείες, σχετικά με την πρόταση οι πολυεθνικές εταιρείες να δηλώνουν τα κέρδη τους, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί σε διεθνές επίπεδο. Στο μια πρέπει να υπάρξει σαφής αναφορά στην επιστημιστική ασφάλεια στα πλαίσια της ε, διαδικασίας ανάπτυξης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το, σε ό,τι αφορά το, το σημείο 41 έχω κάποιες σε κάποια σημεία δεν συμφωνώ. Ο κύριος Ντεζίρ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ζολή για την έκθεσή της και διότι έλαβε υπόψη τις προτάσεις μας παρόλο που εκ νέου υποβάλαμε τροπολογίες ε, αναγνωρίζουμε κάποιες από τις ιδέες μας στην έκθεση που έχει υποβάλει. Ξέρουμε ότι η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και χωρών ΑΚΕ έχει μια ιστορία και ότι θα πρέπει να διατηρήσει αυτόν τον ειδικό χαρακτήρα της χωρίς να ισοπεδωθεί με κάποιους κανόνες όπως αυτούς του ΠΟΕ. Θέλουμε αυτή η εταιρική σχέση παρόλα αυτά να διατηρήσει τη συνοχή όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομικής, εμπορικής, αλλά να λάβει υπόψη και να προωθήσει στόχους όπως ο εκδημοκρατισμός, όπως ε, η πρόθεση και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας όλα τα νέα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας. Η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η μεταφορά τεχνογνωσίας όσον αφορά παραδείγματος χάνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η καταπολέμηση της ε, πείνας, η επισητιστική αυτάρκεια, η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής των φορολογικών παραδείσων. Όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές, επειδή οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης έχουν ε, τεθεί σε ισχύ σταδιακά, κάποιες από τις πρώτες ε, ιδέες και στόχους έχουν πλέον ξεπεραστεί. Θα θέλαμε όμως οι διατάξεις που ισχύουν σήμερα στις χώρες ΑΚΕ να μην είναι λιγότερο πλέον εκτικές για τις χώρες ΑΚΕ, λιγότερο χρήσιμες για τις χώρες ΑΚΕ από αυτές που ίσχυαν στο παρελθόν. Δεν θέλουμε λοιπόν να υποβαθμιστεί η Συμφωνία της Κοτονού. Όσον αφορά την μετανάστευση, θα πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των μεταναστών και να μην υπάρξουν ε, καθεστώτα προς χώρες οι οποίες δεν εγγυώνται τα δικαιώματα των μεταναστών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μισελ, πρόεδρε, επίτροπε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την κυρία Ζολή για την ακρίβεια, την ε, πολύ ε, σαφή και ε, ανάλυση την οποία βλέπουμε σε αυτή την έκθεση η αναθεώρηση της συμφωνίας ε, του Κότονου πρέπει να ενισχύσει τη συμφωνία του Λομέ και τη σχέση μεταξύ των διαφόρων χωρών και η αντιξιακή πολιτική τους πρέπει να εγγυηθεί από αυτή τη συμφωνία. Ο προγραμματισμός, η επανεξέταση και ο έλεγχος της συμφωνίας θα πρέπει να υπαχθούν στην ε, αρμοδιότητα των κοινοβουλίων των ε, στι μας ε, ε, στις χώρες εκεί. πρέπει να ενεργοποιηθούν αυτά τα κοινοβούλια. Αυτή είναι μια προσδοκία την οποία πρέπει να διατυπώσουμε σαφώς στις αρχές των χωρών εταίρων. Ορισμένες κυβερνήσεις δεν προωθούν την κοινοβουλευτική συζήτηση στις χώρες τους όσο θα έπρεπε. Πρέπει επίσης να ενισχυθεί ο δημοκρατικός έλεγχος και ο ρόλος της ισομερούς κοινοβουλευτικής συνέλευσης Ευρω... Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ λαμβάνοντας τις απαραίτητες διατάξεις ώστε οι χώρες ΑΚΕ και να λαμβάνουν τα κείμενα στρατηγικής και περιφερειακής στρατηγικής. Τα περιφερειακά και τοπικά κοινοβούλια πρέπει κατά την άποψή μου να συμμετέχουν πιο ενεργά στη διαδικασία επεξεργασίας των κειμένων εθνικής και περιφερειακής στρατηγικής και μία λέξη για την εργασία της ομερού συνέλευσης πρέπει να έχουμε δύο συνόδους, μία σύνοδος θα εκπέμψει ένα πολύ αρνητικό μήνυμα στις χώρες εταίρους. Πρέπει να οργανώνουμε περιφερειακές συνεδριάσεις πιο τακτικά και στις 25 Ιανουαρίου θα κάνω συγκεκριμένες προτάσεις επ' αυτού στο Προεδρείο της Ισομερούς Συνέλευσης για ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Πρέπει λοιπόν να εγγυηθούμε με πολύ καλύτερο τρόπο την αναπτυξιακή διάσταση όλες αυτές τις προσπάθειες Κύριε Πίτροπε, χαιρετίζω αυτά που είπατε. Υπήρξατε απόλυτα σαφείς ε, για αυτό το θέμα ως επόμενος ε, ε, και επίτροπος εμπορίου είμαι βέβαιος για την, προσπά... για την ειλικρίνειά σας σχετικά με την πρόθεσή σας να δώσετε την δέουσα αναπτυξιακή διάσταση στο... στην όλη αυτή προσπάθεια και θα βοηθήσετε και να δώσετε την απαιτούμενη βοήθεια στις χώρες αυτές για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Ο κύριος Ντέβα για δύο λεπτά. Μιλάμε συνεχώς, ε, μιλάμε για την καταπολέμηση της ένδυας και στην απόπειρα αυτή έχουμε δαπανίσει 350 δις ευρώ περίπου στην καταπολέμηση της ένδυας, ενώ η ένδυα έχει αυξηθεί. Γιατί λοιπόν στις χώρες ΑΚΕ εφαρμόζουμε πολιτικές και προγράμματα που δεν έχουμε καν εφαρμόσουμε στην ίδια ε, την ευρωπαϊκή μας ιστορία. οι Βρυξέλλες δεν έγιναν πλουσιότερες και δεν καταπολέμησαν τη φτώχεια κάνοντας αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς στις χώρες ΑΚΕ. Δημιουργήσαμε πλούτο στην Ευρώπη μέσω δημιουργίας πλούτου. Και πώς δημιουργείται πλούτο στις χώρες ΑΚΕ. Η κυρία Ζολή ε, λέει ότι υπάρχει έλλειψη κεφαλίου. Πολύ ενδιαφέρον. Και επομένως πρέπει ό,τι επενδύουμε σε αυτές τις χώρες να μην βγαίνει. Γιατί δεν χρησιμοποιείται το κεφάλαιο αυτό σε αυτές τις χώρες. Γιατί δεν δημιουργούμε τις προϋποθέσεις προκειμένου το κεφάλαιο αυτό να παραμείνει, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να δημιουργήσει πλούτο. Μέχρι να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτηματικά, κύριε Πρόεδρε, ξοδεύουμε αλόγιστα τα χρήματα των φορολογωμένων μας χωρίς να αποκλείουμε έστω και ένας άνθρωπος να μην είναι πλέον φτωχός. Ευχαριστώ κύριε Ντέβα και για την ε, συντομία σας. Ο κύριος, η κυρία Τζίμερ για δύο, ένα λεπτό. Η πολιτική μου ομάδα στηρίζει την έκθεση της Εύα Ζολή και θα θέλαμε ιδιαίτερα να αναλυφθούν υπόψη κάποια προβλήματα. Όπως τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις χώρες και για τις χώρες και για την κλιματική αλλαγή, η περιφερειακή αντιμετώπιση κάποιων προβλημάτων όσον αφορά τις χώρες ΑΚΕ και την αναπτυξιακή συνεργασία. Η Συμφωνία Κοτονού χρειάζεται να λάβει υπόψη της και τις απαραίτητες επενδύσεις για την υποδομή αλλά και για την στήριξη των κρατικών μηχανισμών. Την ίδια ώρα το θέμα της μετανάστευσης θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις. Με τη συμφωνία της Κοτονού αντιμετωπίστηκε το πολιτικό θέμα της συνεργασίας. Θα πρέπει εδώ να δούμε και το κοινοβουλευτικό θέμα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάθε πενταετία την αναθεώρηση της συμφωνίας αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Με σόκαρε σε μια διάσκεψη επισητιστικής ασφάλειας οι χώρες ΑΚΕ είχαν μια πινακίδα που έλεγε «Μην ταΐσετε την Αφρική, don't feed Africa». Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι η Αφρική δεν χρειάζεται επισητιστική βοήθεια, χρειάζεται επισητιστική αυτάρκεια. Ο πληθυσμός της Αφρικής έχει το ίδιο ενδιαφέρον με τον πληθυσμό στην ε, χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ όπως και στην ε, Νότια Γαλλία. Πρέπει να δοθούν στους αγρότες οι δυνατότητες να αποφασίσουν από μόνοι τους τι πρέπει να παράγουν και να μπορούν να τα πουλήσουν αυτά στις τοπικές αγοράς. Και αυτό είναι προς όφελος του τοπικού πληθυσμού. Να υπάρχει ε, πληθώρα τροφίμων που θα είναι υγιεινή και θα μπορεί να τους βοηθήσει ε, να επιβιώσουν. Η αυτάρκεια λοιπόν, η επισητιστική και η τοπική παραγωγή είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επισητιστική ασφάλεια. Ο κύριος Κάτσμαρεκ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, η δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού έρχεται σε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονική συγκυρία, διότι μπορούμε να επανεξετάσουμε τη Συμφωνία ε, σε ένα ολοένα ε, μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Έγιναν πολλά πράγματα τα δύο τελευταία χρόνια. Είχαμε τη χρηματοπιστωτική κρίση, την αλλαγή του κλίματο, την επιστημιστική κρίση και όλα αυτά φυσικά είχαν επιπτώσει στις αναπτυσσόμενες χώρε. Αυτό που θα έπρεπε όμω να ενδιαφέρει και εμά ε, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο ρόλο τη κοινή κοινοβουλευτική. συνέλευση και το γεγονό ότι θέλετε να μειώσετε τη συχνότητα αυτών των συνεδριάσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο διότι οι χώρες ΑΚΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε καμία περίπτωση δεν συμμετείχαν ε, μέσω της κοινοβουλευτικής του συνέλευσης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών ΑΚΕ. Και πρέπει να δούμε και τι γίνεται με την περιφερειακή διάσταση. Εγώ δεν είμαι κατά της περιφερειοποίησης αυτής καθεαυτής, αλλά πιστεύω ότι δεν θα πρέπει αυτό ε, να υποκαθιστά την κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση. Η κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση θα πρέπει η ίδια να αποφασίζει για τα θέματα που την αφορούν και να μην είναι η συμφωνία αυτή που αποφασίζει. Υποστηρίζω την ε, ε, ανάγκη να ενισχύσουμε τα τοπικά κοινοβούλια. Αναφέρθηκε και κάποιος άλλος στο θέμα αυτό. Στο μέλλον θέλουμε ε, οι χώρε ΑΚΕ να είναι μέλη του Κοινοβουλίου και να μην είναι εκπρόσωποι των κυβερνήσεών του και μόνο, διότι έτσι θα υπάρχει μεγαλύτερη δημοκρατία και επίση θα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή ε, βοήθεια θα μπορούν να αξιολογήσουν τι δραστηριότητε που βοηθούν προ αυτό το στόχο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει πρόσβαση σε έγγραφα στρατηγικού ενδιαφέροντος και φυσικά δεν θα πρέπει να υπάρχει αλληλεοπικάλυψη καθηκόντων. Θα πρέπει να υπάρχει συνέργεση μεταξύ των ε, χωρών και στην κοινή κοινοβουλευτική συνέλευση για να μην υπάρχει... Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το άρθρο 13 της Συμφωνίας του Κοτονού δεν έχει αναθεωρηθεί από το 2000. Αφορά ένα ευαίσθητο θέμα τον διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες ΑΚΕΣ για τα θέματα μετανάστευσης, ισότιμης μεταχείρισης των μεταναστών, τη ρήτρα της μη επαναπρόθεσης, τις βαθύτερες ρίζες της μετανάστευσης και την καταπολέμηση της, το θε... καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και το θέμα της επανεισδοχής, θέματα που ενδιαφέρουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έλλειψη μιας κοινή μεταναστευτικής πολιτικής αντίστοιχη των αξιών της Ευρώπης κινδυνεύει να ενισχύσει στην προβλεπόμενη αναθεώρηση του άρθρου 13 κατασταλτικά μέτρα και την ε, ε, δίωξη των, των ε, παρανόμων μεταναστών. Η σχέση μεταξύ Λιβύης και Ιταλίας που οδήγησε σε παράδειγμα καταστάσεις δεν αποθαρρύνει εκείνους που θέλουν να ενισχύσουν το άρθρο 13 για να υπάρξει ισχυρότερη καταπολέμηση της παράνομης Σε Ορισμένε χώρες το κυνήγι κατά των παρανόμων μεταναστών έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν βεβαίως οι ανησυχίε που δημιουργεί η παρούσα κρίση, αλλά πρέπει να τονίσουμε τη συνέργεια που υπάρχει μεταξύ μετανάστευση και ανάπτυξη. Εάν χρειάζονται βοήθεια οι χώρε ΑΚΕ για την ανάπτυξή του, εμεί χρειαζόμαστε του μετανάστες για να αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση που μας στίζει. Μιλάμε λοιπόν για νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα. Αυτή είναι η τομεί στου οποίου πρέπει να εστιάσουμε τι προσπάθειε μα Είναι τα μόνα στη θέα ασφαλείας για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίσουμε μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρινάλντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ω ε, φιλελεύθεροι δημοκράτε, θέλουμε να δάκραξουμε την ευκαιρία τη δεύτερη αναθεώρησης για να υπάρχει μια ιδέα εξυγχρονισμού, την οποία συμμερίζονται και οι χώρε ΑΚΙΑ. Και όταν μιλάω για εξυγχρονισμό, Μιλάω για πολιτικέ, οι οποίε θα μπορέσουν να επισημάνουν και να επιτρέψουν μεγαλύτερη ελευθερία. Ελευθερία πρωτίστω από την γραφειοκρατία η οποία είναι ολόνα και πιο απαιτητική στις χώρε ΑΚΕ και γίνεται συνεχώς πρόσκομα στην οικονομική ανάπτυξη. Ελευθερία ως δυνατότητα κυρίως για τους φοιτητές για να μπορούν να μεταβούν και να σπουδάσουν στο εξωτερικό και νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε βάσει της αναθεώρησης ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ε, υποτροφιών. Ελευθερία για τις ε, τεχνολογίες ε, πληροφορικές ώστε τουλάχιστον το διαδίκτυο να μπορέσει να γίνει όσο το δυνατόν πιο διαδεδομένο. Και τέλος, ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων προκειμένου να επιλύσουμε και τις ε, μεγάλες ε, παρεμβολές ε, και παραβιάσεις τις οποίες αναφέρθηκε και η συνάδελφος Ντεκέιζερ των συμφωνιών μετανάστευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να βρεθεί σε προεξάρχοντα ρόλο αν μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές. Ευχαριστώ. Νεντελτσέβα για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, καταρχήν συγχαίρω την συνάδελφο, την κυρία Ζολή, για την έκθεσή της. Η αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού θα πρέπει να είναι η στιγμή που θα γίνει ένας απολογισμός και να προταθούν νέες λύσεις όσον αφορά την εφαρμογή και τις συνέπειες αυτής της συμφωνίας. Θα πρέπει να εντοπιστούν οι προτεραιότητες. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και θα αναφέρω τρία σημεία το περιεχόμενο του πολιτικού διαλόγου, γιατί δεν πρέπει που δεν είναι λόγο να χάσουμε από το νου μας τον πρωταρχικό στόχο που είναι η ενίσχυση της ειρήνης, της ανάπτυξης καθώς και η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και ανθρώπινων όντων καθώς και όπλων. Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες αυτών των παράνομων εμπορικών συναλλαγών. Δεύτερον, μια εταιρική σχέση ε, με ευελιξία και με πρωταρχικό στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη η γεωργία, οι θέσεις απασχόλησης για τους νέους, για να νεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να στηριχτούν σε έναν ανοιχτό και δημοκρατικό διάλογο. Τέλος, το θεσμικό πλαίσιο, μια καλύτερη και πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ των αξώνων και των πυλώνων αυτής της συμφωνίας, κάτι το οποίο θα επιτρέψει ένα καλύτερο δημοκρατικό έλεγχο και περισσότερη διαφάνεια. Τελειώνοντα, θα ήθελα να πω ότι κάθε νέο ή αναθεωρημένο εργαλείο θα πρέπει να έχει σαν σκοπό να διατηρηθούν οι στόχοι και το πνεύμα της συμφωνίας. Κεντρικός στόχος είναι η εξάλληψη της πτώχειας και η βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και η σταδιακή ενσωμάτωση των χωρών και στην παγκόσμια οικονομία. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια. Uh, Κύριος Κάσμαν, σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κυρία Ζολή, συγχαρητήρια στον Επίτροπο. Πραγματικά το Κοινοβούλιο θέλει να θέσει στην καρδιά αυτής της συμφωνίας την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και αυστηρές κυρώσεις για τον μη σεβασμό αυτών. Οι διακρίσεις που βασίζονται στο φύλλο, στην αναπηρία, στον σεξουαλικό προσανατολισμό αλλά και διακρίσεις κατά των φορέων του ιού του AIDS είναι απαράδεκτες. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να δούμε ότι καταρχήν υπάρχουν κάποιες υποχωρήσεις που έχουν γίνει και αυτό βασίζεται καταρχήν σε πολιτικές ε, υποχωρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να βάλουμε στην καρδιά τις σχέσεις μας με όλες αυτές τις χώρες και αυτούς τους πρωταρχικούς στόχους και είναι η πρώτη φορά κύριε Επίτροπε, που έρχεστε με αυτό το χαρτοφυλάκιο και παίρνετε το λόγο στο Κοινοβούλιο. Καταρχήν, λοιπόν, θα ήθελα να σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, καθότι πραγματικά είστε πρόσπιστοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα συγχαίρω, λοιπόν, και σα εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα σα θέση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καβάγιο, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Η αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προοδευτική ενσωμάτωση των χωρών και στην παγκόσμια οικονομία. Τα προβλήματα ενεργειακής ασφάλειας, κλιματικής αλλαγής, η παιδεία είναι σημαντικές πτυχές για την ανάπτυξη αυτών των χωρών. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα που χρειάζεται να αντιμετωπιστεί και το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι επίσης ιδιαίτερα ουσιαστικό για την ανάπτυξη αυτών των χωρών ώστε να αποκτήσουν ενεργειακή ανεξαρτησία και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την κρίση που έχει πλήξει τον πλανήτη μας οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν στον τομέα της παιδείας, της κατάρτισης είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας, της μετανάστευσης επιτρέποντας ε, την ε, ενίσχυση της οικονομίας αυτών των χωρών. Θα ολοκληρώσω αναφέροντας τα μικρά, τις μικρές νησιώτικες χώρες οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες λόγω της ιδιαιτερότητάς τους. Η εφαρμογή της Συμφωνίας του Κοτονού πρέπει να λάβει υπόψη αυτό ένα ειδικό σχέδιο δράσης για τις μικρές νησιώτικες χώρες δίνοντάς τους την απαιτούμενη βοήθεια και υποστήριξη για να προχωρήσουν στην βιώσιμη ανάπτυξη. Ο κύριος Φέιο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται ακριβώς αυτή τη στιγμή να πει την άποψή του για τη δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας ε, του Κοτονού. Θα ήθελα να τονίσω τι δυσκολίες αντιμετωπίζονται αυτή τη στιγμή επί του θέματος. Θα ήθελα να ζητήσω να δω τι γίνεται με όλους αυτούς που ζητούν τη βοήθεια της διεθνούς κοινότητας. Ε, σκέφτομαι όλους τους ανθρώπους που ε, έχασαν δικούς τους ανθρώπους και αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρές ε, δυσκολίες. Η Συμφωνία της Κοτονού θέλει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα είναι κοινή αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης από πλευράς χωρών ΑΚΕ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, προάγει την ειρήνη και δημιουργεί ε, ένα δημοκρατικό πλαίσιο συνεργασίας. Η Συμφωνία όταν έγινε έδωσε τη δυνατότητα να γίνουν βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς η πορεία είναι μακρά η χρηματοπιστωτική κρίση, η επισητιστική ασφάλεια, τα θέματα της ενέργειας, ε, το κλιματικό πρόβλημα ε, μας οδηγούν σε μια νέα αναθεώρηση. Και εδώ θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να αυξήσει το επίπεδο της ε, βοήθειάς της ε, στις χώρες ΑΚΕ. Προσυπογράφω την μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινοβουλίων των χωρών αυτών στις μελλοντικέ διαδικασίες αναθεώρησης της συμφωνίας διότι είναι απαραίτητο να συμμετέχουν. Ο κύριος Μάουρο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δεύτερη αναθεώρηση της Συμφωνίας Κοτονού θα πρέπει να έχει ως στόχο να δημιουργηθεί και μια νοοτροπία ευθύνης. Πολύ δύσκολα θα μπορέσει να έχει κάτι τέτοιο χωρίς τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των κρατικών αρχών και των κοινοβουλίων δεν πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να έχουμε πολιτικές οι οποίες θα αντιποκρίνονται εις βάθος στις ανάγκες της ενδιαφερόμενης κοινότητας. Το δεύτερο μεγάλο σημαντικό θέμα είναι η κοινοτική βοήθεια τα 300 δις δολάρια τα οποία δόθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια δεν είχαν καμία επίπτωση αλλά λάβουμε υπόψη ότι η ανάπτυξη της Αφρικανικής Υπήρου στο ίδιο διάστημα ήταν κάτω τους, του 0,2% ετησίω. Είναι αποκαλυπτικό το στοιχείο αυτό και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ξεκινήσει να το λαμβάνει υπόψη αυτό ε, και να αντιμετωπίσει τις αναπτυσσόμενες χώρες ως κοινό τους πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο αφορά σε εμάς την καθημερινή διαβίωση των δικών μας κοινοτήτων. Θα πρέπει καθημερινά με τις τοπικές αρχές να τους βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσουν διότι βρίσκονται και σε μια πορεία νομιμότητας. Και τέλος, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι το να επενδύσουμε σε ανθρώπινο δυναμικό σημαίνει ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονό ότι η μεγαλύτερη επιχείρηση είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από την ένδια. Αυτοί έχουν την ευθύνη να βοηθήσουν την ε, Ήπειρο να ξεφύγει από τον κίνδυνο. Και εμεί έχουμε την ευθύνη να βοηθήσουμε αυτέ τι χώρε με ένα σαφή σκοπό ε, την ευημερία όχι μόνο των χωρών ΑΚΕ, αλλά και των δικών μας χωρών και των δικών μας πολιτών. Θα πρέπει να εστιάσουμε λοιπόν στους ανθρώπους και όχι στα κονδύλια, στην ειλικρίνεια και όχι στα διαφημιστικά μηνύματα. Έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε καλύτερα τις στρατηγικές μας. Η κυρία Ρόιτοβα, 1,5 λεπτό. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για άλλη μια φορά επικρίνω το γεγονός ότι οι αποφάσεις που αφορούν την αναπτυξιακή βοήθεια δεν συμπεριλαμβάνουν ούτε τους μη κυβερνητικού οργανισμούς, ούτε τα κοινοβούλια των κρατών. Δεν έχουμε πρόσβαση στα στρατηγικά πολιτικά έγγραφα. Η Συμφωνία της Κοτονού έγινε ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι δεσμεύσει των κρατών μελών, έτσι ώστε να υπάρξει ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τις χώρες ΑΚΕ, γιατί θα πρέπει και αυτές οι χώρες να έχουν ένα σύστημα διαχείρισης, ένα φορολογικό σύστημα, το οποίο θα μπορεί να καλύψει τους αναπτυξιακούς στόχους. Το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή, τους φορολογικούς παραδείσους και την παράνομη διαφυγή των κεφαλαίων. Σαν αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, θα ήθελα να υπάρχουν τέτοιες διατάξεις στην Συμφωνία Κοτονού. Είναι μια σημαντική ρήτρα που θα πρέπει να συμπεριληφθεί και πολύ λυπάμαι που η έκθεση της ε, κυρίας Ζολή δεν συμπεριλαμβάνει τέτοια ρήτρα. Θα ήθελα λοιπόν η Προεδρία του Συμβουλίου, η Ισπανική Προεδρία, να καλύψει αυτό το κενό. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάει η διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Νίκολας για ένα λεπτό. Επίτροπε, η έκθεση που συζητούμε σήμερα αναφέρεται στην πλήρη ασφάλεια των χωρών ΑΚΕ. Δεν μπορούμε να μιλάμε γι' αυτό χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη κάποιες πραγματικότητες που σχετίζονται ε, με το θέμα της γεωργίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει ρόλο ρυθμιστή στις παγκόσμιες αγορές. Οι εισαγωγές τροφίμων, η αύξηση αυτών των εισαγωγών θα επηρεάσει την, ε, θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των τροφίμων. τα επίπεδα λοιπόν γεωργικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα προς το συμφέρον των χωρών ΑΚΕ και πιστεύω επίσης ότι όλες οι πτυχές της επιστημική ασφάλειας των φτωχοτέρων χωρών σχετίζονται άμεσα με το μέλλον της κοινή αγροτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ κυρία Κύριε Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω την πολύ καλή εκθέση της συναδέλφου, της κυρίας Ζολή. Η εταιρική σχέση μεταξύ χωρών ΑΚΕ και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητη, πιο απαραίτητη παρά Και αυτό μα το δείχνει και η τραγωδία που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στην ΑΕΤ. Μα δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η εταιρική σχέση, η οποία θα πρέπει να ενισχυθεί. Απευθύνομαι στον Επίτροπο, που σήμερα είναι στην ανάπτυξη και αύριο θα αναλάβει τι ε, εμπορικέ συναλλαγέ. Θα σας κάνω τρεις προτάσεις. Πρώτον, να διατηρηθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος με δύο ετήσιες συναντήσεις και όχι μία και ενδεχομένως οι συμφωνίες εταιρική σχέσης να περάσουν από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτών και όχι σε μία απλή εμπορική συμφωνία με τρόπο έτσι ώστε να αναλάβουν τα κοινοβούλια τις ευθύνες τους και τον έλεγχο που πρέπει να ασκήσουν προς όφελος των πληθυσμών. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Φερέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε. Πρόεδρε. Η αναθεώρηση των συμφωνιών Κοτονού θα πρέπει να προάγει τη βελτίωση της πολιτικής συνεργασίας και της ε, αναπτυξιακής βοήθειας. Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και αλληλεγγύη και να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην ε, αυτόνομη ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ. Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί που διατηρούν τις χώρες αυτές σε μια κατάσταση κυριαρχίας. Πολλές φορές υπάρχει ο αυξανόμενος δικός μας ρόλος στη δημιουργία αυτών των σχέσεων. Όσον αφορά τώρα τις ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, οι οποίες ε, βρίσκονται στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, ε, θα πρέπει να αναθεωρηθούν και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη άγουσα. Δεν θα πρέπει να ενισχύσουμε την εξάρτηση των χωρών αυτών από ε, επιχειρήσεις και να είναι όλα προς το συμφέρον των επιχειρήσεων και όχι των λαών. Δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από αυτά οι συμφωνίες ελευθέρων συναναγών. Οι χώρες ΑΚΕ έχουν αποθέματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν σεβαστά και θα πρέπει κάποιο να σεβαστεί και τις θέσεις τους. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κατέργεια να σας πω το σημείο 31 του σχεδίου έκθεσης είναι λογικό και εγώ είμαι κατά των αρνητικών συνεπειών για τους μετανάστες, της υποχώρησης μας όσον αφορά τα δικαιώματα που έχουν σήμερα οι μετανάστες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί. Τέτοιες διεθνείς συμφωνίες έχουν σκοπό να ρυθμίζουν προς όφελος των μεταναστών και των πιο αδύναμων αυτά τα θέματα. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να δώσουμε ένα σωστό μήνυμα, ένα θετικό μήνυμα προς τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι να επιλέξουν σωστές κατευθύνσεις. Έχω επίσης την εντύπωση ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε και την κοινωνική μετανάστευση, κάτι το οποίο μας ε, απασχολεί σήμερα και το οποίο είναι ένα φαινόμενο που θα πρέπει να το εγκαταλείψουμε. Ο κύριος Παπα-Νικολάου. Την συζήτηση για την τεράστια και ασύλληπτη καταστροφή στην ΑΕΤ και το πώς μπορεί η Ευρώπη να συμβάλλει στην ανακούφιση των πληγέντων η συζήτηση αυτή πρέπει να μα υπενθυμίσει και γι' αυτό παίρνω το λόγο σήμερα σε αυτή τη συζήτηση ότι οι συμφωνίες με χώρε που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και που είναι ιδιαίτερα ευάλωτε σε φυσικέ καταστροφέ, όπω απέδειξε η τραγωδία τη Αϊτή, πρέπει να αντιμετωπίζονται από εμά με τελείω διαφορετικό πνεύμα από τι υπόλοιπε οικονομικέ συμφωνίε που συνάπτει η ευρωπαϊκή ένωση. μιλάμε για χώρε όπου μαστίζονται από τη φτώχεια την ανέχεια και τι ασθένειε. μιλάμε για χώρε όπου ο όρο ανθρωπιστική κρίση είναι να γίνει κανόνα. είναι λοιπόν ευθύνη μα, είναι χρέο μα, είναι θεμελιώδη λήθος των πιστεύω μα στην ευρωπαϊκή ένωση όλα αυτά που συζητούσαμε σήμερα και το απόγευμα να βάζουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή και έπειτα τι οποιασδήποτε τεχνικέ και οικονομικέ διαστάσει. για τον λόγο αυτό όλα αυτά που συζητάμε σήμερα τα γραφειοκρατικά ζητήματα τα τεχνικά ζητήματα πρέπει να τα ξεπερνάμε το ταχύτερο δυνατό. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χάνη Πέδρα Μάρτιν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν σκέφτεται κανείς την περιοχή της Καραϊβικής, του έρχονται δύο εικόνες ε, κατά νου. Πρώτον, η σημερινή τεράστια καταστροφή στην ΑΕΤ και αν κάποιος είναι μέλος ε, χρόνια αυτής της κοινοβουλευτικής συνέλευσης θυμάται τις συναντήσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ. Πολλά υπόθηκαν σημαντικά σε αυτές τις κοινοβουλευτικές ε, ισομαρείς ε, συνελεύσεις. Η κατάσταση στην Αιτή όμως, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς τις πολύ πλουσιοπάροχος θα έλεγα, συναντήσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ακία μας και να σκεφτούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο για τις χώρες αυτές και να βοηθήσουμε τις καταστροφές όπως αυτές οι ΑΕΤΗΣ. Πολλά λέμε, αλλά δεν ξέρω αν κάνουμε αυτά που πρέπει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κοινοβουλευτική συνέλευση τη ΑΚΕ είναι πάρα πολύ σημαντική διότι αυτή τη στιγμή η παγκοσμιοποίηση έχει χωρίσει ε, ε, τον κόσμο σε χώρε παραγωγού προϊόντων και σε χώρε προαγωγού ε, προαγωγούς ιδεών. Στο κέντρο αυτή της διαδικασία υπάρχει Μεσόγειος. κόμβο μεταξύ Ευρώπη και χωρών ΑΚΕ. Οι συμφωνίες λοιπόν του Κοτονού θα πρέπει να προσαρμαστούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα και προτείνω ε, και βάσει των όσων είπε ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο Τζόρτζο Ναπολιτάνο, και εγώ να σας πω ότι υποστηρίζω αυτή την πρόταση, θα πρέπει να υπάρχει μία συνέλευση ετησίως της ε, διάσκεψης ΑΚΕ, στην πιο πολυεθνική και πιο μεσογειακή πόλη, την πιο κοντινή στις χώρες ΑΚΕ, την Νάπολη. Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό το ζητά και ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας στις νέες συμφωνίες να μπορέσει να συζητηθεί αυτή η πρόταση. Προσεγγίζεται έτσι η Ευρώπη στους πολίτες και στο λαό της Νότιας Ιταλίας που αποτελεί την πραγματική πλατφόρμα επιμελητίας και προσέγγισης προς τις ε, χώρες της Μεσογείου με τις χώρες ΑΚΕ. Τελευταίος ομιλητής. Πρόεδρε, επέτρεψα στον εαυτό μου να ζητήσει το λόγο μετά από αυτά που είπε ο κύριος Νικουλέσκου, τα οποία θέλω να υποστηρίξω. Στις οικονομικές μας σχέσεις με άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών ΑΚΕ, πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψη την επισητιστική ασφάλεια όπως την νοούμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση διότι έχουμε ορισμένες εμπειρίες. Η μεταρρύθμιση αγοράς της ζάχαρης έγινε σε συνεργασία με τις χώρες ΑΚΕ αλλά δυστυχώς επιδεινώθηκε σαν αποτέλεσμα η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καταστροφική για τους γεωργούς μας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πάντοτε κατά νου την ανάγκη προστασίας επιστικής ασφάλειας της Ευρώπης που χρειαζόμαστε ιδιαίτερα. Ο κύριος Ντεγκούχτ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά το θέμα των του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων, δεν έχουμε καμία αντίρρηση να περιληφθεί στη συμφωνία του Κοτονού, αλλά το, τα συστήματα αυτά είναι μονομερή. Η συμφωνία Κοτονού είναι πολυμερής και γι' αυτό δεν βλέπω πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν στη συμφωνία. Αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τη σχέση δημοκρατικός έλεγχος. Πολλοί ομιλητές ζήτησαν να ενισχυθεί αυτός ο δημοκρατικός έλεγχος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κλήθη να αλλάξει τη θέση της ως προς αυτό το θέμα, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ήδη, αν είναι αυτό δυνατό, οι περιφερειακές συνεδριάσεις να συμπίπτουν με μία από τις δύο ολομέλειες, συνόδους ολομέλειας διότι αλλιώς με όλες τις συνεδριάσεις ε, των, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων θεσμικών οργάνων τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να οργανωθούν. Η ιδέα να έχουμε δύο συνόδους ολομέλειες είναι κάτι με το οποίο συμφωνώ, αλλά θα πρέπει να οργανώσουμε πιο αποτελεσματικά τις περιφερειακές οργανώσεις να λαμβάνουν χώρα περίπου την ίδια εποχή με την Σύνοδο Ολομέλειας. Πολλοί ομιλητές αναφέρθηκαν επίσης στο θέμα των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης. Επ' αυτού έχουμε συμφωνήσει, αλλά ε, αυτό είναι ο όρος πάνω στον οποίο έχουμε συμφωνήσει. Ίσως όμως θα πρέπει να ονομάζονται συμφωνίες ε, εταιρικής σχέσης, ε, αναπτυξιακής εταιρικής σχέσης, για να είναι πιο ανοιχτή η συζήτηση αν το Κοινοβούλιο συμφωνήσει για τη σύνθεση της νέας επιτροπής και είμαι μέλος αυτής της νέας επιτροπής και αναλάβω νέες αρμοδιότητες σε αυτήν θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε οι συμφωνίες αυτές να είναι επιτυχ... να χαρακτηριστούν από επιτυχία, πλήρη επιτυχία. Υπήρξαν επίσης ερωτήσεις για φορολογικά ζητήματα. Νομίζω ότι ήδη απάντησα στην εισαγωγή που σας έκανα. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι σημαντικό αυτό να αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο στις συζητήσεις μα με τις χώρες ΑΚΕ αλλά και στις μεταξύ μας συζητήσεις διότι πρέπει να δούμε με σοβαρότητα το θέμα ξέρω ότι ενδιαφέρεται γι' αυτό και η Ισπανική Προεδρία πιστεύω ότι μπορούμε κάτι να κάνουμε εφόσον βεβαίως έχουμε το σθένος και το θάρρος να συνεργαστούμε με, όλους τους, με όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές και βεβαίως πρέπει να δούμε τι κάνουν οι εταιρείε οι ευρωπαϊκές στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις αναδυόμενες δημοκρατίες και από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχει πρόθεση να ληφθούν σχετικές πρωτοβουλίες. Η μετανάστευση σε ό,τι αφορά το άρθρο 13 και οι δύο πλευρές ε, δέχθηκαν το άρθρο 13 η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, λαμβάνει υπόψη τους τρεις πυλώνες ε, την ανάπτυξη, την παράνομη μετανάστευση και την νόμιμη μετανάστευση και την επανεισδοχή όλα τα σημεία έχουν ληφθεί υπόψη υπόψη, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία θα τηρεί την σωστή ισορροπία ανάμεσα στις, στους τρεις αυτούς πυλώνες. Ο κύριος Κάφμαν είπε κάτι σχετικά με τις διακρίσεις, με τη διακριτική μεταχείριση. Βλέπω ότι δεν είναι πλέον στην αίθουσα ο κύριος Κάφμαν, αλλά έχει απόλυτο δίκιο. Θέλω να πω ο γενετήσιος προσανατολισμός είναι ένα στοιχείο που είχε προταθεί ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε, πρέπει να ξέρουν σε χώρες ε, και απαγορεύεται η ομοφιλοφιλία από τον νόμο. Κάναμε κάποιες παρεμβάσεις σε επίπεδο προέδρων ορισμένων αυτών των χωρών ζητώντας τους να καταργήσουν αυτούς τους νόμους αλλά το θέμα είναι ευαίσθητο και θα χρειαστεί να το αντιμετωπίσουμε το κείμενο είναι σαφές και πιθανότατα δεν θα υπάρξει συμφωνία επ' αυτού αυτή είναι μία δυνατότητα η άλλη δυνατότητα είναι να βρούμε μια διατύπωση η οποία να είναι λιγότερο συγκεκριμένη αλλά να καλύπτει επίσης για το θέμα του γενετήσιου προσανατολισμού. Βεβαίως αυτό είναι κάτι που θα χρειαστεί να συζητηθεί ευρύτερα στο, στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα στα περισσότερα σημεία και ούτως ή άλλως μακρηγόρησα και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Thank you Ευχαριστώ πολύ, κύριε Η κυρία Ζολή για να συνοψίσει εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, από την αρχή της θέσης ισχύ της Συμφωνίας Κοτονού δεν έχει υποχωρήσει η φτώχεια. Δεν μπορέσαμε λοιπόν να ανταποκριθούμε στους στόχους της αποστολής μας. Κάτι πρέπει να αλλάξει με αυτή τη δεύτερη αναθεώρηση. Λοιπόν, είμαι πολύ ευτυχής που διαπιστώνω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη συμφωνία όσον αφορά την υποστήριξη των μέτρων που προτείνω. Και πιστεύω ότι ένα μέτρο που έχουμε στη διάθεσή μας για να δραστηριοποιηθούμε και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε και να εξαλείψουμε τη φτώχεια είναι η καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων. Να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εργαλείο για να είμαστε αποτελεσματικοί στο εσωτερικό λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις χώρες ΑΚΕ μπορούμε να υποχρεώσουμε τις πολυεθνικές εταιρείες να δηλώνουν στην κάθε χώρα που βρίσκονται τα κέρδη τους και τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Πριν όμως αυτό ισχύσει παγκοσμίως θα περάσουν πολλά χρόνια. Ας χρησιμοποιήσουμε σήμερα λοιπόν τις δυνατότητες που μας δίνει αυτή η συμφωνία, τουλάχιστον να εφαρμόσουμε τον κανόνα αυτό στις χώρες μας. Γι' αυτό και σας ζητώ να μην δεχτείτε την τροπολογία που υποβάλλεται για την παράγραφο 16, αλλά να διατηρηθεί η αρχική διατύπωση που ζητά καταρχήν από εμάς τους ίδιους να τακτοποιήσουμε τα πράγματα στις χώρες μας. Επίσης, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να υποχρεώσουμε τις δικές μας τράπεζες επενδύσεων να αποκτήσουν μία δράση κατά των φορολογικών παραδείσων. Θα πρέπει να απαγορεύσουμε τις ε, επενδύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κέρδη στις χώρες τις οποίες είναι εγκατεστημένες, αλλά μεταφέρουν τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους. Αυτό ισχύει παραδείγματο χάρη για την Ζάμπια, ιδιαίτερα για τα 46 εκατομμύρια τα οποία προέρχονται από την εκμετάλλευση ορυχείων, κάτι το οποίο δεν ήταν ωφέλιμο για τον πληθυσμό της χώρας αυτής, αλλά για τους μετόχους της εν λόγω εταιρείας. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να αλλάξουμε τις εντολές που δίνουμε στις επενδυτικές μας τράπεζες και αυτό πρέπει να το κάνουμε τώρα. Υπάρχουν επίσης και κάποιες άλλες αρχές τις οποίες θα πρέπει να υποστηρίξουμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραδείγματος χάρη, τα δικαιώματα των μεταναστών. Και σας ζητώ να διατηρήσετε το άρθρο 31 στην αρχική του διατύπωση και να μην εξαλειφθούν εδώ οι διαμαρτυρίες κατά των διμερών συμφανιών που ουσιαστικά είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ζολή. Σας ευχαριστώ όλους. Τέλος της συνάντησης και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι προφορικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δικονομικά δικαιώματα στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών. Η Βαρόνι Λάτφορντ, καταρχάς,